Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση της κυρίας Μπέρντερ πρόγραμμα δράσης λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας των άγριων ζώων.